Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφέρω ακροθυγώς τα βασικά στοιχεία της αναθεώρησης οικονομικής διακυβερνήσεως που δημοσίευσε